Παρακαλώ λοιπόν όσοι δεν μπορέσατε να κάνετε την επεξήγηση ψήφα, μπορείτε να το κάνετε αύριο ή αλλιώς να τις υποβάλλετε γραπτό.